Catch ούτε μπλε κάρτες. Καλωσορίζω πρώτα απ' όλα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που από ό,τι βλέπω είναι εδώ πέρα σύσσωμη πλην του κυρίου Έτιγκερ. Κάτι λογικό βεβαίως δεδομένης της περίστασης. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για να αιτιολογήσει το αίτημα ο κύριος Τσάνι έχει τον λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. τι προηγούμενε ημέρε, διαβάζοντα τα σχόλια και τι δηλώσει αρκετών συναδέλφων, μου δόθηκε εντύπωση ότι οι περισσότεροι έχουν εκνευριστεί ιδιαίτερω για αυτή την ε, τόσο δυσάρεστη κατάσταση που αφορά τον εκλογέντα κύριο Γιούνκερ. Επομένω, ε, περιμένω μεγάλη υποστήριξη στην πρόταση αυτή, αν και γνωρίζω ότι τα πράγματα θα είναι τελείω διαφορετικά ε, διότι εδώ έχουμε δείξει ότι είμαστε ο ναός της ευρωπαϊκής υποκρισίας. Θα ήθελα να σας κάνω μία, έναν απολογισμό, ξεκινώντας από τους αδέλφους της ΚΟΕ, που δεν ε, φαίνεται να αντιλήφθηκαν ότι πριν από λίγες ημέρες γιορτάσαμε τα 25 χρόνια από την πτώση του τείχους του Βερολίνου και ίσως θα έπρεπε να συνεργαστούν και με αυτούς που θεωρούν ότι δεν θα έπρεπε... Ε, να συνεργαστούν ε, λόγω μιας ε, ε, επίκτητης υπεροψίας. Δεν θα δεχτούμε μαθήματα δημοκρατίας από κανέναν, διότι είδαμε αυτές τις μέρες ποια είναι η δημοκρατία και εμείς να αντιλαμβανόμαστε τελείως διαφορετικά και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Στους πρασίνους θα ήθελα να πω ότι ήγηκε η ώρα να πούνε με ποιους τάσσονται ή με αυτούς που υποκριτικά πρεσβεύουν μια μεγάλη Ευρώπη και ή με αυτούς που θέλουν να την αλλάξουν, δηλαδή εμάς. Μια σαφή επιλογή έκαναν και οι φιλελεύθεροι που με μετά από την ε, συντριπτική ήττα σε ευρωεκλογέ έχουν πλέον ε, συνταχθεί με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και του Σοσιαλιστέ. Από αυτού όμω θα περίμεναν να υπάρχει έστω μια ελάχιστη ένδειξη ε, διότι πραγματικά ο Γιούνκερ έχει καταπατήσει όλα τα ευρωπαϊκά ιδανικά. Θα ήθελα να σταθώ και λίγο στου σοσιαλιστές και στον πρόεδρο Πιτέλα, ο οποίο στις προηγούμενε ημέρε δήλωσε ότι θέλει εξηγήσει από το Γιούνκερ ή αλλιώ θα είχε και αυτός υποστηρίξει την πρόταση μορφή. Έχετε ικανοποιηθεί από τι ε, ε, ανεπαρκείς απαντήσεις του κυρίου Γιούνκερ. Ε, στην πραγματικότητα ε, συμπεριφέρθηκε τελείως διαφορετικά από όσα πρεσβεύει. Εσείς κύριε Πιτέλα ε, αναρωτηθήκατε αν είναι με τους πολίτες ο Γιούνκερ Juncker ή με τους ε, φοροφυγάδες. Ξέρουμε με ποιους τάσεται ο Γιούγκερ και σίγουρα δεν είναι υπέρ των Ευρωπαίων πολιτών, από τους οποίους ως Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου ε, πήρε πάρα πολλά χρήματα για να τα βάλει στις τσέπες των μεγάλων πολυεθνικών. Θεωρώ επίσης ότι ε, δεν θα πρέπει να προασπίζεται τα δικαιώματα των πολιτών. Τα δικαιώματα των πολιτών τα προασπιζόμαστε εμείς που υποτίθεται ότι είμαστε ευρωσκεπτικιστές. Εσείς θέλετε να υπερασπιστείτε τα συμφέροντα των φίλων του Γιούνκερ, δηλαδή των μεγάλων επιχειρήσεων και των ισχυρών δυνάμεων. Πρόεδρε Γιούνκερ, εσείς είστε η χειρότερη εικόνα αυτής της Ευρώπης. Επικεφαλής του Eurogroup υποστηρίξατε όλες τις πολιτικές οι οποίες οδήγησαν στην αποτυχία την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ίδιο καιρό που οδηγούσατε στην Πούλη να την Ελλάδα, εσείς κάνατε συμφωνίες με μεγάλους διεθνείς κολοσσούς. Αν πραγματικά είχατε έστω και ένα ψήγμα αξιοπρέπειας, θα έπρεπε να εσηκωθείτε να φύγετε. Δεν έχετε την αξιοπιστία να εκπροσωπείτε τους Ευρωπαίους και με αυτό το, ε, την πρόταση μομφή ε, θα πρέπει να δείξουμε αυτή την ένδειξη αλλαγή που χρειάζεται η Ευρώπη. Σα δίνουμε τη δυνατότητα λοιπόν να αποδείξετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το μοναδικό νομιμοποιημένο ε, θεσμικό όργανο τη Ευρωπαϊκή Ένωση από του πολίτε, δεν προστατεύει τα δικαιώματα των τραπεζών και των ισχυρών δυνάμεων, αλλά των πολιτών. Σα ευχαριστώ. Äh, Τον λόγο έχει πρώτα απ' όλα εξ ονόματος της Κομισιόν ο κύριος Γιούνκερ. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα ζητώ συγγνώμη για το ότι δεν ε, συμμετείχα εξ αρχής στην συζήτηση. Δεν οφείλεται σε αγένεια, αλλά στο μποτιλιάρισμα μεταξύ Σαβέρνα και Στρασβούργου και ζητώ συγγνώμη για το θέμα της πρότασης Μομφής να πω πως έθεσα και τον εαυτό μου στην διάθεση του Κοινοβουλίου και στις Βρυξέλλες ε, και συζητήσαμε το θέμα αλλά αυτό το οποίο είδαμε στις 13 ε, ε, του μηνός ε, στις Βρυξέλλες και αυτά τα οποία είπα είναι απλά η κατάσταση. Και θα ήθελα να επιστήσω και την προσοχή σε όλους τους συναδέλφους στο γεγονός ότι θεωρώ ότι από αυτή την αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφορετικών ε, νομικών και εθνικών διατάξεων ε, προκύπτουν κάποιες περιπτώσεις οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ακραίες περιπτώσεις και σε αλληλοεπικάλυψη ε, των ευρωπαϊκών θεσμών και έτσι θα είχε χαθεί η ηθική και δεντολογική συνένεση που είναι απαραίτητη για το μέλλον. Επομένως το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο του Λουξεμβούργου, είναι ευρωπαϊκό, διότι οι αποφάσεις αυτές εφαρμόζονται σε 18 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό ακριβώς και πρότεινα και μία σειρά από αλλαγές ε, οι οποίες ε, θα πρέπει να εγκριθούν. Στη διάρκεια της προεκλογικής ε, εκστρατείας, ε, στις 15 Ιουλίου, όταν ανέλαβα ε, τα ηνία, όταν ανέλαβα τα ηνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επίσης τον Οκτώβριο, επέμεινα για την δημιουργία ενός συστήματος, ώστε να υπάρχει και μία βάση κοινή φορολογική για τις επιχειρήσεις. Ε, είπα ότι είμαι υπέρ του φόρου για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, ότι πλέον ε, δεν είναι θέμα με αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά επειδή έχει ξεκινήσει μια διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας, ε, αφορά συγκεκριμένα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή. Και επίσης ζήτησα να υπάρχουν και κάποιες συνεργασίες μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης φορολογικές πολιτικές. στο Brisbane, στην Αυστραλία, ε, υποστήριξα υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης το G20 ε, της ε, Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας και εκεί διαπίστωσα ότι το G20 δεν ήθελε να συμπεριλάβει στα συμπεράσματά του την απαραίτητη αναφορά στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τη διαφάνεια σε θέματα φορολογικών αποφάσεων. Ε, όλοι οι Ευρωπαίοι θα το είχαν υποστηρίξει. Εκτό και αν αυτοί οι οποίοι δεν εξέφρασαν την άποψή του, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν διαφορετική άποψη, γι' αυτό και δεν μίλησαν. Θα ήθελα επίση να επιστήσω και την προσοχή σα στο γεγονό ότι όταν ε, το 2005 είχαμε την ε, Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευρά Λουξεμβούργου, είχα προτείνει στο ΕΚΟΦΗΝ να υπάρχει μια φορολογική αρχή ε, που να είναι τελείω διαφορετική από την Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή για να μπορούμε να παρακολουθήσουμε και την εφαρμογή των συμπερασμάτων ε, ε, του Eurogroup ε, και τον κανόνα, τους κανόνες διοντολογίας που είχαμε εγκρίνει στη διάρκεια της Προεδρίας μου. Όλα αυτά βέβαια δεν οδήγησαν σε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Είχα ζητήσει από το Συμβούλιο την Ιταλική Προεδρία να ξαναπροτείνει στο Συμβούλιο Εκοφίλ και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τη δημιουργία μιας επιτροπής, φορολογικής επιτροπής που θα έχει ακριβώς τα καθήκοντα αυτά και να προετοιμάζει τις αποφάσεις και, ε, όπως κάνει και η Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή και προετοιμάζει τα, ε, τις αποφάσεις για το ΕΚΟΦΗΝ. Και ναι, μενει η πρόταση μορφή ε, γίνεται βάση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά θα προτιμούσα να είχε γίνει σε μια πιο κατάλληλη στιγμή, ε, μετά το τέλο Νοεμβρίου, να έρθω εδώ να σα μιλήσω και Βλέποντα την ταυτότητα των ε, όσων υπογράφουν αυτή την πρόταση μομφή, πραγματικά αναρωτιόμαι ποια ήταν τα κίνητρά του. Ε, κάθε φορά βέβαια που θα μου το ζητάτε θα απαντώ στις ερωτήσεις που μου θέτετε, αλλά έχω την εντύπωση ότι οι προθέσεις ε, των όσων συνέταξαν αυτή την πρόταση μομφής δεν είναι αυτές ε, οι οποίες μας είπαν, διότι ότι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εγώ δεν είμαι φίλος των μεγάλων κεφαλαίων, και ορισμένες φορές ε, υπήρξαν και κάποιες πολυεθνικές οι οποίες ε, δεν μπόρεσαν να κάνουν απρόσκοπτα αυτό που θέλουν, όπως με κατηγορείτε. Να σας πω το εξής. Η πρόταση μορφή αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και έχω την εντύπωση ότι ε, μόνο εμένα ουσιαστικά θέλετε να κατηγορήσετε. Λέω λοιπόν, είπα εδώ ενώπιον του Κοινοβουλίου στις 15 Ιουλίου ότι εάν ποτέ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποσύρει την εμπιστοσύνη του σε ένα μέρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το συγκεκριμένο μέλος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα κληθεί να παραιτηθεί. Ε, ε αφήστε ησύχου λοιπόν στους υπόλοιπους επιτρόπους. Αν θέλετε να φύγετε, να φύγω, πέστε το και θα φύγω. Σας ευχαριστώ κύριε Γιούνκερ. Ξεκινάμε τώρα με την συζήτηση για το ΕΛΚ. Τον λόγο έχει ο πρόεδρος, ο κύριος Βέμπερ. Κύριε πρόεδρε, κύριε πρόεδρε της Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα το συζητήσαμε στην προηγούμενη Ολομέλεια στις Βρυξέλλες. Ο κύριος Γιούνκερ αναφέρθηκε στο θέμα της φορολογικής δικαιοσύνης στην Ευρώπη και το τι θέλει να κάνει και εμείς πράγματι θέλουμε να σταματήσει αυτή η πρακτική των μεγάλων ομίλων ε, που μπορούν να μην πληρώνουν φόρους αλλά θέλουμε ε, για να προχωρήσει αυτό το θέμα χρειαζόμαστε μια επιτροπή η οποία θα επιδείξει κάποια πρωτοβουλία. Γι' αυτό έχει την πλήρη στήριξή μας ε, ο κύριος Γιούνκερ και η επιτροπή του και την Πέμπτη θα καταψηφίσουμε το το ότι βρίσκεται εδώ πέρα σύσσωμη επιτροπή είναι πραγματικά σημαντικό μήνυμα ότι θέλουν να δουλέψουν και θέλουμε εμείς να τους στηρίξουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Φαράτζ, Λεπέν και οι λοιποί που υπέγραψαν έχουν τώρα ξανά τα δύο λεπτά δημοσιότητας ε, στα ΜΜΕ αλλά θα ήθελα να σα υπενθυμίζω πως όλοι οι βουλευτές εδώ πέρα έχουν τα ίδια δικαιώματα. Όχι, κατα... όταν κατατίθεται ένα αίτημα το συζητάμε και θα ψηφιστεί. Αλλά ποτέ δεν εργάζεστε επικοδομητικά, μόνο καταστροφικά. Και ειλικρινά, ειλικρινά σας λέω, με τη σημερινή συζήτηση σκέφτομαι πως για το θέμα το οποίο μιλάμε σήμερα ε, είναι ιδεώδες υποτίθεται για εσάς κύριοι κύριε Φαράτζ και κυρία Λεπέν. Δεν έχει αρμοδιότητα η Ευρώπη, κανένας επίτροπος, κανένας κακός γραφειοκράτης της Βρυξέλλες. Είναι στα χέρια των κυρίαρχων κρατών μελών, όπως ακριβώς το θέλετε, όπως είναι τα ιδεώδη σας. Και πρακτικά ερωτώ, γιατί δεν δουλεύει τότε, γιατί δεν λύνεται το πρόβλημα στον ιδεώδη κόσμο που ζει ο κύριος Φάραντς και η κυρία Λεπέν. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρώπη που έχετε εσείς κατά νου είναι αυτό ακριβώς το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει. Κύριε Φαράτζ, εσείς φταίτε που δεν πληρώνουν οι μεγάλοι όμιλοι φόρους. Γιατί δεν υπάρχει ακριβώς καμία συμφωνία για αυτό το θέμα. Και μια που μιλάμε για την ομάδα EFTT. Κοιτάξτε την ομάδα αυτή. Ο κύριος Τσάνι από την ομάδα του κυρίου Γκρίλο. Λέτε εμείς είμαστε η Ευρώπη. Αναρωτιέμαι δηλαδή όταν λέτε εμείς είμαστε η Ευρώπη ποιοι είστε ακριβώς. Γιατί ε, οι μεν του Γκρίλο λένε θέμε αλληλεγγύη με τη μετανάστευση. Ο κύριος Φάρατς μας λέει ότι θα πετάξει και τους Ρουμάνους έξω. Υπάρχουν εντωμεταξύ Ρουμάνοι και Πολωνοί στην ομάδα σας που λένε θέλουμε τα ίδια δικαιώματα και εμεί με τις ε, παλαιές χώρες. Και ταυτόχρονα η κυρία Λεπέν λέει δεν θέλω εγώ αλληλεγγύη σε αυτή την Ήπειρο. Ε, έχετε λοιπόν πολλές ε, ομάδες ε, εδώ πέρα που είναι κατά των προσφύγων, κατά των ξένων, κατά των Εβραίων γενικώ. Αυτή είναι η νέα Ευρώπη που θέλετε να μας παρουσιάσετε. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είστε η νέα Ευρώπη, είστε η παλιά Ευρώπη. Κύριε Πρόεδρε. Εγώ χαίρομαι για την ψηφοφορία της Πέμπτης. Εγώ θέλω να συνεχίσει να εργάζεται η Κομισιόν. Θα δούμε τώρα από αυτή την ψηφοφορία εάν θα σημειώσουν μία νίκη οι λαϊκιστές και οι ακροδεξιοί. Εγώ δεν θέλω να συμβεί κάτι τέτοιο. Τον λόγο τώρα για τους ε, σοσιαλδημοκράτες έχει ο πρόεδρος, ο κύριος Πιτέλα. Κύριε Πρόεδρε, μου φαίνεται λίγο σουρεαλιστικό το γεγονός ότι η παρουσίαση μιας πρότασης μομφής, αντί να μας εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους κατατίθεται η πρόταση, είναι απλώς ένας οριμαγδόν προσβολών κατά ε, πολιτικών ομάδων και ευρωβουλευτέ που το μόνο του ελάττωμα είναι ότι σκέφτονται λογικά και μπορούν και θέλουν να αποφασίσουν για μια πρόταση μορφή αν θέλουν να την υπερψηφίσουν ή να την καταψηφίσουν σε σχέση με τα συγκεκριμένα πράγματα που προτείνονται. Εγώ συνήθως δεν απαντώ σε προσβολές. Διότι υπάρχει ένας παλιός κανόνας που λέει ότι όποιος φτύνει στον αέρα θα τον πετύχει στο κεφάλι αλλά υπάρχει κάτι το οποίο αξίζει της απάντησής μου. Και είναι η κατηγορία εδώ στην αίθουσα, διότι κοιτάξτε εδώ έχουμε εκατοντάδες συναδέλφους, άνδρες και γυναίκες που συχνά διαφωνούν. Αλλά πάντα, πάντα υπερασπίστηκαν την αξιοπρέπεια και το κύρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό υπερεθνικό όργανο το οποίο εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες και εμείς εδώ εκπροσωπούμε εκατομμύρια πολίτες. Ωστόσο, με την πρόταση μομφής, Καλό θα ήταν να έχετε καλή αγωγή, γιατί ο πρώτος κανόνας είναι οι καλοί τρόποι. Εγώ δεν απάντησα στον συνάδελφο όταν επιτέθηκε στην ομάδα μου και σε μένα και εσείς πραγματικά είστε αγενείς. Τίποτα άλλο. Με τη σημερινή πρόταση μορφής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να μπει στην ιστορία. Δεν νομίζω ότι έχει συμβεί ποτέ να υπάρχει πρόταση μορφής ε, κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 24 ημέρες αμέσως μετά την, ε, το διορισμό της. Να δούμε τι θα συνέβαινε εάν στέλναμε σπίτι τους όλους τους επιτρόπους. Το πρόγραμμα επενδύσεων των 300 δισεκατομμυρίων, το οποίο θα ανακοινωθεί σε δύο μέρες, θα τυναζόταν στον αέρα. Θα διαγράψουμε έτσι την τελευταία ευκαιρία της Ευρώπης να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να αντιμετωπίσει την κρίση. Θα ξεκινήσουν ε, ε, διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων μεταξύ των κρατών μελών για τον διορισμό της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα αφιερώσουμε μήνες για να συσταθεί μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και στο μεταξύ θα καταρρεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν θα υπάρχουν απαντήσεις, θα εκτοξευθεί η ανεργία και η πυρός μας θα βρεθεί σε αποπληθωρισμό. Αυτό θέλετε. Αυτό πραγματικά θέλετε. Να μείνουμε σε αυτή την κατάσταση, να μην υπάρχει καμία απάντηση. Αυτό είναι αυτό που ζητάτε. Εμείς λοιπόν δεν το δεχόμαστε. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί Επίτροποι, αυτό το οποίο θα πρέπει να φοβάστε σήμερα είναι η πρόταση μομφή των πολιτών εάν δεν κάνουμε τίποτα για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Θα μα πετάξουν όλου έξω. Όλου. Και εγώ λοιπόν σα λέω, στρωθείτε στη δουλειά προκειμένου να ξεκινήσει το σχέδιο των επενδύσεων, να καταπολύσουμε τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή και τις πρακτικές των πολυεθνικών οι οποίες φοροδιαφεύγουν και φοροαποφεύγουν με ε, τη συνενοχή πολλών ε, κυβερνήσεων. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και εμείς ε, σας ρωτήσαμε πριν από δύο εβδομάδες κύριε Πρόεδρε από αυτού και μας είπατε ότι θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να εναρμονιστούν τα φορολογικά μας συστήματα και μας πείσατε στο περιεχόμενο, στην ουσία. Εμείς δεν σας δώσαμε μια δήλωση, σας δώσαμε εμπιστοσύνη βάσει της ουσίας των προτάσεών σας. Και γι' αυτό ακριβώς θα επαγρυπνούμε. Δεν ξυπνάμε τώρα δεν ε, θέλουμε να περιμένουμε να βγουν επιχείρη οι τίτλοι στις εφημερίδες για να καταγγείλουμε φορολογικές πρακτικές των πολυεθνικών και των κυβερνήσεων. Το Κοινοβούλιο εργάστηκε. Α υπενθύμισα κάποιε προτάσει οι οποίε περιλαμβάνονται σε έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε στην προηγούμενη θητεία, που είναι πολύ συγκεκριμένε προτάσει, τι οποίε εμεί θα ε, τι εμπιστευτούμε στο έργο της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό είναι ο σοβαρός τρόπος για να καταπολεμήσουμε τη μεγάλη μάστιγα της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγή. Αλλά αυτό είναι και ο σοβαρός τρόπος για να μπορέσει να προχωρήσει μία κυβέρνηση, μία επιτροπή και ένα Ευρωπαίος πρόεδρο, για να μπορέσουν να εργαστούν διότι εργάζονται προ όφελο των συμπολιτών μα. Για την ομάδα ECR, ο κύριος Λεγκούτκο έχει το λόγο. Uh, Ευχαριστώ. Δεν θα μιλήσω για προσωπικές αρετές και λατώματα των εμπνευστών του ψηφίσματος. Τους γνωρίζω. Ούτε περί των προθέσεων γιατί δεν με αφορούν, δεν με ενδιαφέρουν. Θα μιλήσω για το πρόβλημα Juncker. Υπάρχει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, να σας πω. Πρόεδρε, δεν ξεκινάτε καλά. Ας το ομολογήσουμε. Και εγώ δεν είμαι ικανοποιημένο μετά όσα είπατε την περασμένη φορά. Ούτε μας πείσετε με, τα, με τις σημερινές δηλώσεις. Να το πω αλλιώς δεν νομίζω ότι έχετε και την παραμικρή τύψη. Σπάνιο βεβαίως μεταξύ πολιτικών αν και όχι αδύνατων. Κάτι όμως πρέπει να είναι σαφές. Χρειαζόμαστε πλήρη εις βάθος ενημέρωση για τις φορολογικές συμφωνίες και όλε όλες τους τις προεκτάσεις. Το χρειαζόμαστε. Εμείς, οι Ευρωπαίοι λαοί, οι λαοί της Ευρώπης, οι λαοί οι οποίοι έχασαν δισεκατομμύρια λόγω αυτής της ανήθικης πονηριάς των ηγετών του Λουξεμβούργου. Δεν είναι αμεληταίο το θέμα. Όταν λέω λοιπόν εμείς, ενώ επίσης οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η πλειοψηφία των οποίων σας υπερψήφισε προσφάτως κύριε Γιούνκερ. Πρόεδρε Γιούνκερ, θα ήταν καλό και για σας. Γιατί ό,τι και να κάνετε ως πρόεδρος της Κομισιόν, η σκιά αυτού του σκανδάλου θα σας ακολουθεί με το όνομά σας γραμμένο επάνω της. Έως ότου το θέμα ξεκαθαριστεί πλήρως και μια για πάντα. Και ποιος πρέπει να διεκπαιρέωσει αυτήν την έρευνα, εννοείται οι αρχές του Λουξεμβούργου κατά κύριο λόγο, αλλά και ανεξάρτητες αρχές, διεθνείς αρχές όπως όσα. Είμαι όμως ανήσυχος παρόλα αυτά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με εσάς πρότεινε στο τιμόνι και όντας υπεύθυνο για την έρευνα. Εγώ προσωπικώς είμαι προσχολημενο στο νεμό Ιουντέξιν Καμσασούα. Κανείς δηλαδή δεν μπορεί να δικάζει τα δικά του πράγματα, τις δικές του υποθέσεις. Κανείς δεν μπορεί να είναι κριτής των δικών του υποθέσεων. Αυτή η αρχή του ρωμαϊκού δικαίου δεν μπορεί να παραβιαστεί εκτός αν θέλουμε να αυτογελιοποιηθούμε. Θα ήταν κάτι απαράδεκτο. Όπως θα ήταν επίσης απαράδεκτο να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ευκαιρία για να ενημερώσουμε την φορολογική νομοθεσία στην κατάσταση που είναι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό τη δική σας ηγεσία, Πρόεδρε Γιούνκερ. Για τους φιλελεύθερους, ο Πρόεδρος, ο κύριος Φερχόφστατ. Πρόεδρε, εγώ προσωπικώς πιστεύω ότι δεν πρέπει να σπαταλήσουμε πολλά λόγια επί του ψηφίσματος. Γιατί? Διότι όλοι αισθάνονται, διαισθάνονται ακόμη και οι εκπρόσωπος της ECR ότι εδώ παίζεται ένα παιχνίδι από δύο ομάδες την Ευρώπη Ελευθερίας και η Δημοκρατίας, τον κύριο Φάρατζ και την ομάδα της κυρίας Λεπέν. Το καταλαβαίνω αυτό το παιχνίδι. Είναι φυσικό. Έτσι γίνεται στην πολιτική. Πρόκειται για μια διεστραμμένη όμως λογική. Περί αυτού πρόκειται. Τι θέλουν οι δύο ομάδες να κρίνουμε επί του LuxLeaks των διαρών αυτών πριν καν αποφανθούν οι αρμόδιες αρχές. Ε, δεν είναι σοβαρό αυτό. Να καταθέσουμε ένα ψήφισμα δηλαδή τη στιγμή ακριβώς που ζητήσαμε από την Κομισιόν να εντρυφήσει τα ζητήματα αυτά και πριν καν συστήσουμε μια κοινοβουλευτική επιτροπή διερεύνησης. Δεν θα ήταν λοιπόν ανοησία να ξεκινήσουμε κάτι τέτοιο πριν καν ξεκινήσουμε τη διαδικασία διερεύνησης. Πρόεδρε, για μένα το μόνο ενδιαφέρον αυτού του ψηφίσματος, δεν είναι το περιεχόμενο, είναι το γεγονός ότι εν τέλει ο κύριος Φάραζος και η κυρία Λεπέν αποκαλύπτουν την κρυφή του σχέση. Αυτό είναι το σημαντικό και αυτό είναι το ενδιαφέρον αυτού του ψηφίσματος. Αυτό που έκρυβαν λοιπόν τόσον καιρό. Γιατί έκρυβαν ότι έχουν την ίδια στρατηγική. Αυτά δεν λέει ο κ. Φάρετζ στου ε, ψηφοφόρου του. Είναι απόδειξη λοιπόν ότι το UKIP είναι ένα ρατσιστικό, αποτρόπαιο, ξενόφοβο κόμμα και δεν λίγο έχω κι άλλα να σας πω. Ένα Ισλαμόφοβο κόμμα. Και αυτά δεν είναι δικά μου λόγια. Είναι τα λόγια του ιδρυτή του UKIP, του Αλασκάτ. Κατά τη γνώμη μου, το λέω προς τον κύριο Ζάνη, εδώ το διακύβευμα δεν είναι η αποφυγή φόρων. Άλλο είναι το παιχνίδι. Ο κύριο Ζάνη ε, δείχνει προς εμάς, κατηγορεί εμάς πριν τακτοποιήσει τα του οίκου του. Ο κύριος Φάραντς θα έπρεπε να δει τα του οίκου του. Ο ίδιος το Isle of Man, στην ίσο του Man, έχει παράκτη, έξω Και το λέω και προς την κυρία Λεπέν διότι σε λίγα λεπτά θα γίνουμε θύμερα της οργής της κυρίας Λεπέν, η οποία δανείζεται από ρωσικές τράπεζες για να χρηματοδοτήσει την πολιτική της δράση και κανείς δεν εξανίσταται περί αυτού. Πιστεύω λοιπόν, και το είπε και ο κύριος ε, Φέμπερ, μίλησε τη γλώσσα της αλήθειας, ότι εσείς κύριε Φαράτζ και οι ομοίοι σας είστε κατά της Ευρώπης. Μην νομίζετε λοιπόν ότι με τον τρόπο αυτό θα καταρακώσει την Ευρώπη. Η απάντησή μου είναι απλή. Ας επιστρέψουμε λοιπόν στη δουλειά μας και σήμερα ας καταψηφίσουμε αυτό το ανόητο ψήφισμα. Παρακαλώ. Μα κύριε Πρόεδρε, θεωρείτε πως αυτός ο σχορός λόγος ενισχύει την αξιοπιστία του Κοινοβουλίου ή όχι. εξαιώματο τη Καλώς τον λόγο έχει η κυρία Τσίμερ εξ ονόματος της Ενωμένης Αριστεράς. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Γιούνκερ, η κριτική μας στο πρόσωπό σας εξακολουθεί να υφίσταται την ασκήσαμε και στις ακροάσεις και όταν ήρθατε στην ομάδα μας και τότε είχαμε πει πόσο προβληματικό είναι κατά την άποψή μας το ότι το Λουξεμβούργο είναι φορολογικός παράδεισος για τις επιχειρήσεις και ακριβώς να εμφανίζεστε και να μας λέτε πως θέλετε να κλείσετε αυτά τα παραθυράκια και να φροντίσετε για δίκαιη φορολογία όταν έγιναν γνωστά τα έγγραφα και μιλάμε εδώ πέρα μόνο για έγγραφα επιχειρήσεων που συνεργάζονται με την ε, PricewaterhouseCoopers. Μόνο από αυτούς ε, μιλάμε για 340, 340 επιχειρήσεις οι οποίες ε, έλαβαν εκατοντάδες αποφάσεις όπως τις λέγατε από τις εφοριακές αρχές του Λουξεμβούργου προς το συμφέρον τους. Και ξεκαθαρίσαμε πώς θα πρέπει από εδώ και μπρος η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάει προς περισσότερη αλληλεγγύη, προς μια χρηματοδότηση μιας αλληλέγγυας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αυτός είναι ο δρόμος της αξιοπιστία. και σας ρωτήσαμε ποια ήταν η δική σας άποψη και μπορώ να πω εξ ονόματος της ομάδας μου. Απογοητευτήκαμε και από την ομιλία σας πριν από 10 μέρες. Περιμέναμε κάτι ξεκάθαρο. Περιμέναμε να καταλάβετε πως δεν είναι μόνο προσωπική η κριτική σε εσά. Είναι κριτική σε ένα σύστημα το οποίο πλέον φέρει το όνομά σας, το σύστημα Juncker. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι προσωπικό δικό σας, γιατί είπατε παρενθετικά πως 22 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ακριβώς αυτό το ίδιο σύστημα. Ρωτήστε τον κύριο Φερχόφστατ και του υπενθυμίσατε το δικό του ρόλο. Δικαίως. Αλλά το θέμα εδώ πέρα, όταν μιλάμε για αξιοπιστία, αυτό το οποίο θα περιμέναμε ήταν να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Εσείς προσπαθήσατε να μας πείτε πως ε, ως πρόεδρος της Κομισιόν δεν θα μας μιλάτε για τα του Λουξεμβούργου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν το δεχόμαστε. Και τότε εμείς προσπαθήσαμε να υποβάλουμε πρόταση μομφής, δεν μαζέψαμε τις υπογραφές. Γιατί δεν θέλουμε εμείς υπογραφές από τους ακροδεξιούς εθνικιστές γιατί η Ευρώπη που θέλουν αυτοί οι βουλευτές είναι μια διαφορετική Ευρώπη. Και ζητήσατε να αλλάξετε την Ευρώπη μαζί μας. Ναι, αλλά προς τα πού θα πάει αυτή η αλλαγή. Αυτό είναι το βασικό. Και ακριβώς αυτό διακρίνει το δικό μας το ψήσιμο και το δικό μας το αίτημα από το δικό τους. Αν δηλαδή είχαμε κοινό αίτημα με τον κύριο Φάρατς και την κυρία Λεπέν, ε, δεν γίνεται. Όχι, δεν, δεν μπορούμε να συνυπογράψουμε μαζί τους. Εσείς λοιπόν πρέπει να πείτε θέμε να αλλάξουμε, πρέπει να υπάρξει μια αλληλέγγυα κοινωνική Ευρώπη. Αλλά πρέπει να αποφασίσετε κι εσείς με ποιον θα είστε, με ποια ομάδα θα είστε. Εμείς και είμαστε και απογοητευμένοι από τους πράσινους, το λέμε, και τους σοσιαλδημοκράτες, γιατί πριν από 10 μέρες δεν εκμεταλλευτήκατε την ευκαιρία μαζί μας να συζητήσουμε το θέμα και να γίνει εδώ πέρα η συζήτηση. Ποια άλλη Ευρώπη θέλουμε στο θέμα το φορολογικό. Ήταν ευκαιρία. Τώρα έχουμε την ευκαιρία τουλάχιστον να γίνει μια διερευνητική επιτροπή. Έχω 4,5 λεπτά. Α, α συγγνώμη μια εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή που είναι περισσότερο από ε, την επιτροπή που θα συσταθεί τώρα. Πρέπει λοιπόν να σταματήσει τουλάχιστον η πρακτική που ακολουθείται μέχρι τώρα. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, εδώ μόλις ακούστηκε μία από τις πιο σοβαρές κατηγορίες που θα μπορούσε να ακουστεί. 24 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποκαλέστηκαν ρατσιστές. Και εγώ δεν μπορώ να φανταστώ κάτι πιο σοβαρό. Αυτό παραβιάζει το άρθρο 11 που λέει ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα σέβονται ο ένας τον άλλον βάσει ε, των αρχών που καθορίζονται στον κανονισμό. Όταν υπάρχει λοιπόν παραβίαση τέτοιας μορφής, κύριε Πρόεδρε, το άρθρο 165 και το 166 ε, καλεί τον Πρόεδρο να ανακαλέσει ε, τον Ευρωβουλευτή στην τάξη. Και εσείς δεν κάνετε τίποτα. Γιατί? Σας ευχαριστώ κύριε Βουλευτά. Δεν, με, δεν μπορώ ξανά εντύπωση ότι ξέρετε αυτά τα άρθρα πολύ καλά. Η δηλώση του κυρίου Φερχόστατ ήταν ε, τσιτάτο δήλωσης του ιδρυτού του UKIP. Δεν άκουσα κάτι το οποίο να απευθύνεται προς τον κύριο Φαράτζη ή κάποιον άλλον. Επιτρέπεται νομίζω να μεταφέρουμε τα όσα είπε ο ιδρυτής του κόμματός σας εντός της αιθούσης. Η κυρία Χάρμς μετά, μετά την ε, κυρία Χάρμς. Κυρίες και κύριοι, κύριε Γιούνκερ, κυρίες και κύριοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα των Lux Leaks για να το αφήσουμε σε αυτούς που κάθονται σε αυτή την πτέρυγα των, ε, της ε, αίθουσας. Τώρα, εντάξει δεν ξέρω μπορεί να κάνω λάθος για το κίνημα των πέντε αστέρων, αλλά ας το αφήσουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε, το θέμα μας απασχολεί γιατί η δημοσίευση των Lux Leaks ήρθε ακριβώς στη στιγμή στην οποία θέλαμε να κάνουμε μια νέα αρχή με περισσότερη αλληλέγγυα πολιτική. Και πράγματι αυτό το οποίο κάνει το LuxLeaks είναι να δημιουργεί νέα μεγάλη δυσαρέσκεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποδεικνύει ότι η βασική αρχή της Ευρώπης δεν είναι η αλληλεγγύη, αλλά ο καθένας προσπαθεί να υποβεληθεί εις βάρος των άλλων και κοιτάει την πάρτη του πώς φτάσαμε ως εδώ είναι ένα ζήτημα, αλλά αυτή είναι η αντίληψη πολλών ανθρώπων, ειδικά στις χώρες στις οποίες φροντίσαμε με την πολιτική λιτότητα να μην λειτουργούν πλέον τα κράτη όπως θέλουν οι άνθρωποι και οι μικρές επιχειρήσεις που πληρώνουν τους φόρους τους και αναμένουν να λειτουργούν τα κράτη. Γι' αυτό εγώ αναμένω η συζήτηση για το ποια είναι τα έσοδα που χρειάζονται τα κράτη για να λειτουργούν προς όφελος των πολιτών τους είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει. Και αν ο κύριος Τσάνι τώρα θεωρεί πως εγώ ανήκω στο, στους εκπροσώπους του μεγάλου κεφαλαίου, τι να πω. Θέλουμε να ξεκαθαρίσει αυτό το ζήτημα ανεφόρον και θεωρούμε πως δεν θα γίνει τώρα αυτό ακολουθώντας τη γνωστή αυτή η ερωτελεστία φέρτε μου την κεφαλή του Ζαν Κλοντ και μετά όλα θα γυρίσουν στην παλιά κατάσταση. Αντιθέτως εμείς θεωρούμε πως ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ ακριβώς γιατί είναι αυτός τον οποίον κοιτάει αυτή τη στιγμή όλη η Ευρώπη και έχει απαιτήσει και προσδοκίες από αυτόν, ο κύριος Γιούνκερ θα αλλάξει ακριβώς τα πράγματα στο Λουξεμβούργο και σε άλλες χώρες, στην Ολλανδία, στην Ιρλανδία, στην Αυστρία, όλα αυτά τα οποία είναι στραβά με την ανοχή όλων των ε, Πρωθυπουργών και Υπουργών Οικονομικών. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ξεκαθάρισμα της υπόθεσης αυτής για να βγάλουμε ακριβώς τα διδάγματα τα οποία πρέπει. Να τελειώσει επιτέλους αυτή η αιώνια διαφωνία για μια κοινή φορολογική βάση. Και πλέον εδώ πέρα κύριε Γιούνκερ το ζήτημα είναι υπαρξιακό. Είτε θα το ξεκαθαρίσετε, ξέρω πως δεν μπορείτε να το κάνετε μόνο σας, είτε όμως θα το καταφέρετε εσείς με το ευρωπαϊκό πνεύμα το οποίο έχετε επιδείξει. Ή πραγματικά τα πράγματα θα γίνουν πολύ σκοτεινά. Και δεν είναι, απευθύνομαι εδώ πέρα σε ολόκληρη την Κομισιόν, δεν είναι το πρόβλημα μόνο του κυρίου Γιούνκερ. Το θέμα είναι ακριβώς αν θα έχουμε μια επιτυχημένη θητεία της Κομισιόν ή δεν θα γίνει τίποτα στο τέλος. Γιατί η εμπιστοσύνη των πολιτών είναι αυτό το οποίο έχει πληγεί. Σας ευχαριστώ. Επί της διαδικασίας ε, και ο Σκάβα έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συνεχίσω από τον συνάδελφο. Νομίζω ότι είναι σαφές, ανεξάρτητα από τις απόψεις ε, του καθενός εδώ στο Κοινοβούλιο, υπήρχε σαφής ε, κατηγορία από πλευρά ε, των όσων ακούστηκαν από τον κύριο Φερχόφστατ. Και παρακαλώ κοιτάξτε τον κανονισμό. Ήταν πολύ σοβαρέ οι κατηγορίε και ισχυρισμοί και ο κύριο Φερχόφστατ θα ήθελε να ρωτήσει τον συνάδελφο, τον κύριο Μπεσέρ που κάθεται εδώ δίπλα μου, αν είναι κατά των Ισλαμιστών. Κατά του Ισλάμ, μάλλον. Okay. Μάλιστα. Συνεχίζουμε για την ομάδα ευθυντή, ο κύριος Γούλφ. Κύριε Γιούνκερ, πρόκειται για σκάνδαλο, ένα φορολογικό σκάνδαλο το οποίο δεν εξατμίζεται. Η απάτη έχει παρισφρήσει εκεί ακριβώς που κάθεστε και όσο κάθεστε εκεί η ατμόσφαιρα θα γίνεται όλο και χειρότερη. Σήμερα εσείς είπατε εδώ ότι δεν είστε φίλος του μεγάλου κεφαλαίου. Κι όμω ήσασταν επικεφαλή του Λουξεμβούργου, ήσασταν πρωθυπουργό και επιτρέψατε σε εκατοντάδε πολυεθνικέ να συνεργαστούν με τι φορολογικέ αρχέ και να αποφύγουν φόρου. Αν αυτό δεν είναι είμαι φίλο των επιχειρήσεων, των μεγάλων επιχειρήσεων, τι είναι. Κάποιε τέτοιε επιχειρήσει πλήρωναν 1% φόρο. Και τώρα μα λέτε ότι είστε αλληλέγγυο με του λαού τη Ευρώπη. Ναι, το πιστέψαμε, οι λαοί της Ευρώπης, αυτοί που πληρώνουν το τίμημα της λιτότητας, της φτώχειας, η οποία σαρώνει την Ευρώπη ως πάλι πανούκλα. Και εσείς φροντίζετε να αποφαληθούν αυτοί οι λαοί από τις δικές σας απάτες. Η Γερμανία, η Αγγλία, η Γαλλία, η Ιταλία δεν είδαν να έχουν τέτοιες συμφωνίες και κάποιε εταιρείε να πληρώνουν 1% φόρο. Μιλήσατε για αλλαγή συμπεριφορά. Πιανού συμπεριφορά. Η μόνη συμπεριφορά που πρέπει να αλλάξει είναι η δική σα. Και ζητάτε από άλλου σε αυτό το κοινοβούλιο να μην σα επιτίθενται. Πού ήταν όμω η δική σα αλληλεγγύη όταν επιβάλλετε μια τρόικα στην Ελλάδα. Όταν εσεί ταυτόχρονα στο Λουξεμβούργο απαλλάσσετε από του φόρου από εκατομμύρια τι πολυεθνικέ εταιρείε. Τι κάνετε για την Ιταλία με την ανεργία του 55%. Τι έκανε το Λουξεμβούργο λοιπόν όταν υπέγραφε αυτέ τι συμφωνίε εξ ονόματο υποτίθεται τη Ευρώπη. Αναδοηθείτε είστε όντω οι θεματοφύλακε τη ηθική εξ ονόματο των ανθρώπων που σα ψήφισαν. Ή μήπω φροντίζετε για τον εαυτούλη σα. Πιστεύω ότι κάθε τόσο έρχεται η στιγμή να παλαστεί σώμεθα από αυτούς οι οποίοι δεν πιστεύουν στο ευρωπαϊκό ιδεώδες το οποίο εμείς οι άλλοι πιστεύουμε. Ευχαριστώ. Das Wort hat jetzt die Abgeordnete Λόγο έχει κυρία Λεπέν. Κύριε Πιτέλα, ξεχνάτε στην αποκαλυπτική σας ε, παρέβαση, Ξεχάσατε την εισβολή των ακρίδων και επιτεθήκατε κι εσείς ε, μαζικά με ένα λεξιλόγιο το οποίο δυστυχώς ε, είναι απίστευτο. Στην πραγματικότητα, χάρη στη διαρροή των εγγράφων, πιστήκαμε για την απάντηση στο Λουξεμβούργο. Πάνω από 300 πολυθυνικές υπέγραψαν με τις φορολογικές αρχές συμφωνίες για να εξασφαλίσουν εκπτώσεις στους φόρους τους. Και τα κέρδη μετά επανέρχονται στο Λουξεμβούργο μέσω διαφόρων τεχνασμάτων. Αυτά γίνονταν σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εις βάρος και της Γαλλίας. Χάρη στον κύριο Γιούνκερ, οι δικέ μα τώρα εταιρείε ακριβώ πληρώνουν περισσότερα, επειδή κάποιε δικέ του εταιρείε πληρώνουν λιγότερα δεν είναι μόνο του Λουξεμβούργο σε αυτό, αλλά είναι πρωταθλητής. Έχουμε διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιεί το Λουξεμβούργο. Συνεργασία μεταξύ θηγατρικών, πολυεθνικών, μεταφορά κερδών, ενδομπηλικές συναλλαγές, έτσι για να μην πληρώνει τελικά κανείς φόρο. εντοπίσαμε τέτοιες τεχνικές, τέτοιες τακτικές, μειωμένο ΦΠΑ για παράδειγμα, ώστε κάποιες επιχειρήσεις να μπορούν να πουλάνε στη Γαλλία πληρώνοντας λιγότερο φόρο στο Λουξεμβούργο. Πρόκειται για μια φορολογική απάτη. αξιοποιώντας τους κανόνες, παρεβιάζοντας τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χάρη σε φοροτεχνικούς και συμβούλους που πληρώνονται αμύθιτα ποσά. Κύριε Γιούνκερ, ο του του παλιός υπουργό μας, έλεγε πριν καιρό στην Γαλλική Γερουσία ότι το Λουξεμβούργο είναι αλληλέγγυο το πρωί και το βράδυ κλέβει από τις τσέπες μας. Κύριε Γιούνκερ, είσαστε 100% υπεύθυνο. Εσείς θεσπίσετε όλους αυτούς τους κανόνες, δώσατε τη δυνατότητα σε αυτές τις πολυεθνικές να κάνουν αυτά που έκαναν. Δεν είστε ειλικρινείς και δεν πιστεύουμε ότι μπορείτε να δώσετε μάχη για να ανατρέψετε αυτά τα οποία κάνατε. Θα ήταν σαν να βάζουμε τον Αλ Καπόνε, πρόεδρο τη Επιτροπής Ασφάλειας. Γι' αυτό λοιπόν υποστηρίζουμε το ψήφισμα αυτό και ζητούμε από όλου τους πολιτικούς που θέλουν να δώσουν τη μάχη κατά τη φοροαποφυγή να καταψηφίσουν την Επιτροπή Juncker. Βεβαίω, δεν είστε ο μόνο, επαναλαμβάνω, είστε όμω το καλύτερο παράδειγμα σε αυτήν την τακτική. Εμείς σας υπερψηφίσαμε όμως. Το ΕΛΚ, οι σοσιαλιστές, οι φιλελεύθεροι, αυτοί σας υπερψήφισαν και αυτοί σας έβαλαν εκεί που είστε. Σύμβολο δηλαδή της ε, απάτης, της διαφθοράς, σύμβολο της υποστήριξης των μεγάλων επιχειρήσεων που κερδοσκοπούν εις βάρος των φτωχών. Παρακαλώ κύριε Γιούγκερ. Κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ μεγάλη η πρόκληση να απαντήσω μόνο στην κυρία Λεπέν, η οποία κάθε φορά που παίρνει το λόγο με γεμίζει ε, γλυκόλογα εδώ στο ημικύκλιο. Αλλά πέραν αυτού θα ήθελα να απαντήσω και σε κάποια στοιχεία τα οποία προέκυψαν από τη συζήτηση. Κυρία Τσίμερ, μιλήσατε για σύστημα Juncker. Με ποιο δικαίωμα. Εσείς και πολλοί άλλοι συνάδελφοι μιλήσατε για το σύστημα που υποτίθεται ότι φέρει το όνομά μου, το οποίο είναι το αποτέλεσμα διαφόρων διατάξεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σας παρακαλώ μην δίνετε στο σύστημα αυτό το όνομά μου, ένα σύστημα το οποίο δεν ξεκίνησα εγώ, δεν ε, βοήθησα εγώ. Είναι απλά διάφορες διατάξεις διαφόρων κρατών. Είπα ενώπιόν σας, επαναλαμβάνοντας ότι η Επιτροπή της οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω θα καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή και τη φοροφυγή. Το είπα εδώ ενώπιόν σας πριν από 15 ημέρες με ποια μέσα θα προσπαθήσουμε τα αποτελέσματα αυτά της ε, φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής να μην επαναληφθούν, ε, της μη φορολόγησης και φυσικά και από δεντολογικό και ηθικό επίπεδο. Ζήτησα από τον συνάδελφο τον κύριο Μοσκοβισή να ετοιμάσει μια οδηγία η οποία θα ε, προβλέπει την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση φορολογικών θεμάτων μεταξύ των 28 κρατών μελών. Και φυσικά ε, θα ήθελα όλες οι πολιτικές ομάδες ε, να υποστηρίξουν αυτή την άποψη. Κανείς δεν είπε ότι δεν θέλει να γίνει κάτι τέτοιο, όπως πραγματικά θέλω να πιστέψω ότι και στις χώρες σας, τα κόμματά σας, τα εθνικά σας κοινοβούλιο θα κάνετε ό,τι μπορείτε ώστε τα 28 κράτη-μέλη να βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή την ε, προσπάθεια. Βασίζομαι σε εσά. Δεν χρειάζεται να κάνω τώρα παθητικές εκκλήσεις. Πραγματικά θα πρέπει να φροντίσουμε σε κάθε χώρα να υπάρχει συνένεση γύρω από αυτή την ιδέα σε θέματα ε, προληπτικών φορολογικών αποφάσεων και να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών αυτόματα. Στο Brisbane στην Αυστραλία όταν πρότεινα το συγκεκριμένο κανόνα και είπα ότι θα πρέπει να γίνει παγκόσμιο κανόνας, είδα ότι ε, ήταν πολύ ε, μετριοπαθής ο ενθουσιασμό των υπολείπων και επομένως θα πρέπει εμείς να φροντίσουμε να υπάρξει συνένεση με βάση αυτή την ιδέα όλες οι πολιτικές ομάδες, όλα τα μέλη εδώ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, αν κατάλαβα καλά, θέλουν να με υποστηρίξουν όταν ζήτησα από την Ιταλική Προεδρία και από τη μελλοντική φυσικά Προεδρία να συστήσει μια φορολογική ομάδα στο Συμβούλιο Υπουργών και στα κράτη-μέλη, ώστε να υπάρχει αυστηρή εφαρμογή των απαιτήσεων που προκύπτουν από τον κώδικα δεοντολογίας ε, ε, για τα φορολογικά ζητήματα, το οποίο καθορίσαμε το 1997. Κανεί δεν το αρνήθηκε αυτό και σήμερα διαπιστώνω ότι όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμφωνούν ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ε, ισότιμο όργανο με την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων που θα φροντίζει να υπάρχει κατάλληλη εφαρμογή των φορολογικών κανόνων και φυσικά θα βοηθά και το Συμβούλιο Υπουργών όταν θα πρέπει να απαντήσουν και να αποφασίσουν επί του συστήματος και ζητώ να υπάρχει φορολογική εναρμόνιση. Κάτι το οποίο φυσικά δεν θα πρέπει να είναι εις βάρος της, ε, του φορολογικού ανταγωνισμού. Όταν είναι αθέμητος ο φορολογικός ανταγωνισμός ε, είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσει να καταπολεμήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με όλες τις, τις δυνάμεις. Και φυσικά δεν θα πρέπει να αμφισβητείτε τα λεγόμενά μου. Μιλώ ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μιλώ ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώπιον του οποίου δεσμεύομαι εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να φροντίσουμε ένα από τα ουσιαστικά στοιχεία του προγράμματος του οποίου σας παρουσίασα και βάσει του οποίου εξελέγην, ε, είναι το θέμα αυτό. Ε, εγώ θα το τηρήσω και όλοι οι Ευρωπαίοι Επιτροποί θα προσπαθήσουν να το τηρήσουν και όλοι όσοι υποστήριξαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της οποίας προεδρεύω θα φροντίσουν το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να, εφαρμοστεί καταρχήν και σε όλες τις λεπτομέρειες. Και ε, γι' αυτό δεσμεύτηκα. Έχω ένα συμβόλαιο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εξελέγει με βάση αυτό του προγράμματο, βάση του προγράμματο των επενδύσεων των 300 δισεκατομμυρίων που θα σα παρουσιάσω την Τετάρτη ε, το πρωί εξελέγει με βάση ε, συγκεκριμένες αρχές που αφορούν ε, όχι μόνο τα θεμέλια της δημοκρατίας αλλά και συγκεκριμένους φορολογικούς κανόνες που είπε ότι θα εφαρμόσω και πραγματικά πρέπει να σας πω ότι όλοι όσοι γνωρίζουν το ζήτημα και είναι και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν διατελέσει πρωθυπουργοί, υπουργοί οικονομικών με υποστήριξαν σε αυτή την κίνηση και σας το λέω με πάσα σοβαρότητα. Ακούστε σταματήστε να με προσβάλλετε. Εντάξει, εγώ προσβάλλομαι. Υπάρχουν κάποιοι εδώ μέσα που δεν θίγονται καν. Έκανα αυτό το οποίο υποσχέθηκα και θα το κάνω στο 100% των δυνάμεών μου. Σας ευχαριστώ. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε ψηφοφορία την 5η το μεσημέρι στις 12 η ώρα. Συνεχίζουμε με τη μερίσια διάταξη.